Okay, ξεκινήσουμε γιατί έχουμε καθυστερήσει κιόλας. Ε, καθυστερήσαμε με τους συντονιστές και είμαι σίγουρος πως τα μέλη θέλουν να προχωρήσουμε γρήγορα στην ψηφοφορία. Είμαστε στο σημείο 7 ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία και ανταλλαγή απόψεων επί του σχεδίου έκθεσης. Η συγητής είναι ο Εντουάρντ Σικλού, να έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Νομίζω οι στατιστικές ανέκαθεν ανέκαθεν είχαν να κάνουν με αριθμητικά στοιχεία και απηχούσαν αυτά που θεωρητικά έπρεπε να απηχούν και μετά όλα συνεχίζονταν ε, κανονικά. Όμως σήμερα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και τον κίνδυνο που αφορά την έλλειψη αξιοπιστίας στις ίδιες τις στατιστικές. Την έλλειψη εμπιστοσύνης δηλαδή. Αυτό στο παρελθόν έχει να κάνει με στοιχεία των ε, κρατικών δημοσιονομικών. Όμως πρόσφατα Είχαμε και άλλο πρόβλημα με στατιστικά δεδομένα, το ίδιο το Λίμπορ. Όλοι θεώρησαν ότι αυτό είναι δεδομένο και τελικά έχουμε βρεθεί με, αντιμέτωπο με το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Ναι, πολύ μεγάλα προβλήματα. Εκατοντάδες τρισεκατομμύρια δολάρια παραγόγων προϊόντων βασίστηκαν σε έναν δείκτη που όλοι μπορούσαν να μετατρέπουν ανάλογα με το πώς ε, τους βόλευε. Η έκθεση αυτή λοιπόν είναι εξαιρετικά επίκαιρη. Υπογραμμίζει τις απαιτήσει ποιότητας. Απαιτούμε υψηλή ποιότητα για τα στατιστικά μας δεδομένα. Τα όργανα οικονομικής πολιτικής και τα ίδια αποτελέσματα έχουν πληγεί ακριβώς από την έλλειψη εμπιστοσύνης, αξιοπιστίας και τη χαμηλή ποιότητα των στατιστικών δεδομένων. Τα στατιστικά στοιχεία θα πρέπει να είναι αξιόπιστα για το κοινό, όπως και τα θεσμικά όργανα και ο αλληλοσυσχετισμό τους. Όταν προκείται ένα τέτοιο σκάνδαλο, τα ίδια τα θεσμικά όργανα πλήττονται. Τα τραπεζικά ιδρύματα, χάνουν την αξιοπιστία τους ως αποτέλεσμα τέτοιων ε, καταστάσεων και σκανδάλων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε αυτή την πραγματικότητα και στο παρελθόν δημοσίευσε το έγγραφο αυτό για μια δυναμική διαχείριση της ποιότητας. Έχουμε και εμείς μια δική μας, πρωτοβουλία, έκθεση μας πρωτοβουλίας έκθεσης για το ίδιο θέμα και τώρα έχουμε και την νομοθετική έκθεση ενώπιον μας. Η ίδια η έκθεση θέλει να δώσει έμφαση στο ότι δεσμεύσεις εμπιστοσύνης θα πρέπει να αφορούν και τις κυβερνήσεις που να αναλάβουν ενεργά το ρόλο τους και να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των επίσημων στατιστικών δεδομένων με το σεβασμό της ανεξαρτησίας των εθνικών στατιστικολογικών, στατιστικών μάλλον, Ινστιτούτων. Χρειαζόμαστε διαφανείς διαδικασίες πρόσληψης, βασιζόμενοι μόνο σε κριτήρια επαγγελματικών προσόντων. Η πρόταση απαιτεί αναθεώρηση του υπάρχοντος βασικού νομοθετικού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές και τα ευρωπαϊκά στατιστικά δεδομένα, ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη αξιοπιστία. Πιο συγκεκριμένα, η επαγγελματική ανεξαρτησία των εθνικών στατιστικών αρχών είναι άκρα σημασία σε αυτό το επίπεδο. Η υπάρχουσα πρόταση αναφέρεται στους επικεφαλείς των εθνικών στατιστικών ιδρυμάτων ως ε, επαγγελματιών που πρέπει να φέρουν εις πέρα στα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία ώστε να εξασφαλίζουν το κύρος του ίδιου του ιδρύματος στο οποίο εργάζονται. Είναι απαραίτητο να έχουν την ελευθερία να αποφασίζουν για τις διαδικασίες και τις μεθόδους και θα πρέπει να τους απαγορεύεται να αναζητούν και να λαμβάνουν οδηγίες από εθνικές κυβερνήσεις. Αυτό είναι καθοριστικό για να υπάρχει ανεξαρτησία την οποία επιζητούμε. Θα πρέπει να υπάρχουν διαφανείς και νομικώς δεσμευτικοί κανόνες για τον διορισμό, την ε, μεταφορά ή την απόλυση σε ιδρύματα και υψηλότερου επίπεδου, όπως και οι τράπεζες πολλές φορές γνωρίζουν. Θα πρέπει να υπάρχει αιτήσια έκθεση για τις στατιστικές ε, δραστηριότητες και τη δημοσιονομική κατάσταση από την ε, εν λόγω αρχή και αυτές θα πρέπει να είναι στο δυνατόν διαφανέστερες. Θα πρέπει να, να γίνει σεβαστός ο κώδικας πρακτικής των τατιστικών ιδρυμάτων από το 2009, αλλά σύμφωνα με την πρότασή μας θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι εδώ θα προσυπογράψουν οι κυβερνήσει όλων των κρατών μελών. Και επίση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η δέσμευση αυτή θα γίνει σεβαστή. Υπάρχει το νέο άρθρο 17α για την πρόσβαση στη χρήση και την ένταξη των ε, διοικητικών στοιχείων. Ο πρωταρχικό στόχο εδώ είναι να καταρτιστεί ένα νομικό πλαίσιο για την ε, εντατική χρήση των δημοσιονομικών, δημόσιων μάλλον πόρων, για την κατάρτιση των ευρωπαϊκών δεδομένων, στατιστικών δεδομένων. Και στο άρθρο 6 υπάρχει μια τροπολογία για να διασφαλίσουμε την ανεξάρτητη θέση τη Eurostat τη ίδια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ολοκληρώνω λέγοντας ότι δεν απαιτείται να υπάρξουν εδώ πρόσθετοι πόροι για τα κονδύλια των στατιστικών στοιχείων. Απλώς πρέπει να βελτιωθεί ο συντονισμός και η συνεργασία. Ενώ ταυτόχρονα να διασφαλιστεί υψηλότερη ποιότητα για τις ίδιες τις στατιστικές. Σας ευχαριστώ. Okay, um shadows. Ωραία, περνάμε στους ε, σκιώδεις εισηγητές. Ο Ζαν Πολ δεν είναι εδώ. Ε, είναι... Η Ρόδη, εσείς είστε η σκιώδη εισηγητρία, ωραία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον εισηγητή που έρχεται με συμπληρωματικές πληροφορίες και προτάσεις, ένα θέμα που πράγματι μας έχει απασχολήσει στο παρελθόν, διότι όλη η προσπάθεια, όχι μόνο για την αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων και των αρχών που τα εκδίδουν, άρα και των χωρών που έχουν την ευθύνη να τα προμηθεύουν στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία είναι άμεσα συνδεδεμένο με αυτές τις αλλαγές και τις δεσμεύσεις, τις νομικές δεσμεύσεις που πρέπει να πετύχουμε. Παράλληλα όμως δεν είναι μόνο θέμα αξιοπιστίας, είναι και ένα θέμα ε, καλής λειτουργίας του νέου συστήματος δημοσιονομικού ελέγχου, ε, συγκρίσιμων στοιχείων, ε, αξιολόγησης της πρόοδου των κρατών μελών και επίτευξης μιας ε, ε, οικονομικής ε, συνοχής και συντονισμού των οικονομικών πολιτικών. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό θέμα αυτό που συζητούμε σήμερα, διότι χωρίς αξιόπιστα και ενδολεχή στοιχεία στατιστικά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ούτε στην αποτύπωση της πραγματικότητας ούτε στο συντονισμό των κρατών μελών. Λοιπόν, υποστηρίζουμε τις, τις προτάσεις του εισηγητή ε, γιατί πρέπει αφενός να είμαστε σίγουροι για την ανεξαρτησία των αρχών που εκδίδουν τα στατιστικά στοιχεία. Πρέπει όμως ε, παράλληλα να είμαστε και σίγουροι για την ε, βάση αυτών των δεδομένων και για την συγκρισιμότητα μεταξύ των χωρών μελών. Είναι λοιπόν γεγονός ότι η νέα προσπάθεια για παρακολούθηση της, του συντονισμού των δημοσιονομικών και οικονομικών πολιτικών, όλες οι δεσμεύσεις ε, που έχει πάρει η Επιτροπή μας, ε, το Κοινοβούλιο μας, βασίζονται σε καλά αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με τους τρόπους συλλογή, την ανεξαρτησία και την ε, αξιοπιστία των αρχών που τα εκδίδουν. Και θα δούμε στη συνέχεια πώς θα συμπληρώσουμε αυτή την πρόταση με επιμέρους ιδέες της πολιτικής μας ομάδας. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, Σε ευχαριστώ, Σοφή. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Νομίζω πως οι προτάσεις αυτές είναι πράγματι πολύ χρήσιμες, αλλά έχω κάποιες ερωτήσεις, όχι πολλές. Η πρώτη μου ερώτηση είναι εάν τα ίδια κριτήρια θα ισχύσουν και για τον διορισμό του διευθυντή της Eurostat. Τα ίδια κριτήρια ανεξαρτησίας. Δεύτερον, για τις λεγόμενες δεσμεύσεις για την εμπιστοσύνη στα στατιστικά στοιχεία. Τι να σας πω, εμένα μοιάζει σαν υπόσχεση στην ε, προσκοπική μας τιμή. Ε, θα έπρεπε να έχουμε κάτι πιο δεσμευτικό Ειδικά αν δούμε πως κάποιοι από τους μη δεσμευτικού ε, κανόνες ε, που υιοθήθηκαν ε, τα προηγούμενα χρόνια δεν γίνονται σεβαστοί από τα κράτη-μέλη. Και αυτή είναι η αίσθηση που έχω γενικώ. Ακούμε πολλά πράγματα για τα στατιστικά στοιχεία τα τελευταία χρόνια και κάθε φορά φαίνονται τα πράγματα καλά στα χαρτιά, αλλά ξέρουμε πως η πράξη είναι διαφορετική. Πώς θα έπρεπε λοιπόν να δούμε και τον τρόπο επιβολής είναι ένας κύριος εδώ πέρα μπροστά μου, αν μπορεί να περιμένει λίγο μέχρι να τελειώσω. Yes. Ε, με συγχωρείτε, συγγνώμη. Έχασα τον ήρμό μου τώρα. Και τέλος, θα ήθελα να μου εξηγήσετε τι εννοείται εδώ πέρα με την πλήρη πρόσβαση σε όλα τα διοικητικά έγγραφα πώς θα ερμηνευτεί αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Φιλίπ. Ακούστε, θεωρώ πως έχουμε μια καλή βασική πρόταση από την ε, Κομισιόν και είναι μια καλή βάση για τη δουλειά μας. Θέλω να κάνω κάποια σχόλια. Πρώτα απ' όλα για αυτό το οποίο είπατε, Εντουαρτ, για το ότι οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες πρέπει να είναι ανεξάρτητες. Ε, ως προς τον καθορισμό της μεθοδολογίας. Ναι, μπορώ να συμφωνήσω σε ένα βαθμό, αλλά ας δεχτούμε και το ότι πως ειδικά όταν μιλάμε για στατιστικά στοιχεία η μεθοδολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο να ορίσουμε το ποια τελέσματα θα έχουμε. Δεν υπάρχει, όπως ξέρετε, ουδέτερο στοιχείο και οι άνθρωποι οποίοι στελεχώνουν τις στατιστικές υπηρεσίες δεν είναι ρομπότ, είναι άνθρωποι με ιδέες, ε, με πιστεύω. Και όπως δεν θέλουμε να εμπιστευτούμε ε, ένα κεντρικό τραπεζίτη να είναι τελείως ανεξέλεγκτος, δεν θεωρώ πως θα πρέπει να δώσουμε πλήρη ε, ελευθερία σε μια στατιστική υπηρεσία να χρησιμοποιήσουν όποια μεθοδολογία θέλουν. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ πως ο νομοθέτης έχει ρόλο να παίξει δίνοντας μια κατεύθυνση για το τι, σε τι είδου ε, τομείς θέλουμε δεδομένα. Θυμάμαι την όλη συζήτηση που είχαμε στο εξαπλό πακέτο για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Είναι νομίζω πολιτική επιλογή να ορίσουμε ποιου δείκτες θέλουμε να παρακολουθούμε και πιθανώς να μαζεύουμε και ε, ποια δεδομένα θα έχουμε και αν αφήσουμε αυτές τις επιλογές ε, μη ερετούς ε, και ανεξέλεγκτους αξιωματούχους πού θα καταλήξουμε, θα έχουμε την ίδια κατάσταση. Δηλαδή, και εγώ μπορώ να πω, όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι πράσινοι. Ναι, δηλαδή θέλω να είναι ανεξάρτητοι, αλλά μία κατεύθυνση πρέπει να είναι ε, θέμα της πολιτικής εξουσίας και οπωσδήποτε των κοινοβουλίων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Όσον αφορά τώρα τους εθνικούς κώδικες ε, πρακτικής, βεβαίως πρέπει να είναι κατανοητή για το μέσο πολίτη και επίσης θέλουμε να επιβάλλονται. Με άλλα λόγια δηλαδή, Ούτως ή άλλως και με τις τράπεζες δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την αυτορύθμιση, δεν θα είμαστε λοιπόν ικανοποιημένοι και με την αυτορύθμιση αυτών των υπηρεσιών. Εάν υπάρχει κώδικα συμπεριφορά, πρέπει να είναι δεσμευτικός και αναλόγως να εφαρμόζεται. Επίσης κάτι το οποίο πρέπει να δούμε είναι το πώς μπορούμε να προωθήσουμε την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να έχουμε κάποιον ε, μηχανισμό ελέγχου από τους ε, ομολόγους τους και τέλος είμαστε ικανοποιημένοι από τον τωρινό ρυθμό ανταλλαγής ε, στοιχείων μεταξύ Eurostat και Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών. Εγώ δεν είμαι προσωπικά ικανοποιημένος. Ε, μάλλον σε αυτά τα σημεία θα καταθέσουμε τροπολογίες. Ευχαριστώ Βίκη. Ευχαριστώ. Όπως θα γνωρίζουν και οι συνάδελφοι, συμφωνώ απολύτως με τις εκκλήσεις για περισσότερη διαφάνεια και μεγαλύτερη ανεξαρτησία των πληροφοριών για τους πολίτες, τους φορολογουμένους, τους ε, ψηφοφόρους μας και τους δικαιούχους των κονδυλίων. Η ανεξαρτησία είναι καθοριστική σημασία εδώ. Δεν θα πρέπει να υπάρχει πολιτική παρέμβαση ούτε για τις προθεσμίες όταν οι πληροφορίες δημοσιεύονται, για το πότε δηλαδή θα δημοσιοποιηθούν και πρέπει να υπάρχει ανεξαρτησία αλλά και υψηλή ποιότητα. Όχι ανεξαρτησία και χαμηλότερη ποιότητα. Νομίζω τα σχόλια που έχουν κάνει ως τώρα τα, οι συνάδελφοι για τα ίδια τα πρότυπα που θέλουμε να θέσουμε είναι πολύ σημαντικά. Συμφωνώ απολύτως με τη Σόφη ότι η διατύπωση στο κείμενο για την πρόσβαση σε όλα τα διοικητικά αρχεία τι ακριβώς εννοούμε εδώ Πιανού τα αρχεία. Ποια είναι τα αρχεία που θα ζητώνται. Είναι λίγο ευρία, λίγο ε, πλατιάζει αυτή η φράση. Πολλές φορές έχουμε πει σε συναντήσεις μας ότι για επιχειρήσεις θα πρέπει να μπορεί να απαιτείται να προσφέρουν τις ίδιες πληροφορίες με διαφορετικούς μορφότυπους και να μπορούν αυτές οι πληροφορίες να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά. Αλλά αν τώρα λέμε ότι οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες μπορούν να πηγαίνουν και να ξεφυλίζουν τα αρχαία όλων των διοικητικών υπηρεσιών, εδώ θα πρέπει να συνεχίσουμε καλύτερα τι εννοούμε. Νομίζω ότι υπάρχει λοιπόν περιθώριο να δουλέψουμε πολύ περισσότερο το ιστορικό αυτής της πρότασης για να βεβαιωθούμε ότι θα θέσουμε σωστούς στόχους ανεξαρτησίας και υψηλής ποιότητας, χωρίς όμως να ξεπερνούμε τα διαχωριστικά για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών και προκειμένου να έχουμε αποτελεσματική χρήση των πληροφοριών υπάρχουν και δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κόστος και τον έλεγχό του. Δεν θέλουν να υπάρξει μεγαλύτερος ε, φόρτος και κόστος για την κοινωνία. Αυτό είναι φυσικά λογικότατο και είναι η σωστή κατεύθυνση, σωστά την δεικνύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έγιναν επίσης και σχόλια για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, καμιά φορά, όπως λέμε, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειε αλλά είναι και ένα ζήτημα το τι θέλουν και τι δεν θέλουν να αποκαλύπτουν τα κράτη-μέλη. Εδώ θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσο το θέμα αυτό θα λάβει και σοβαρέ πολιτικέ διαστάσει. Θα πρέπει να είμαστε λεπτομερεί και συγκεκριμένοι στο τι θέλουμε να εκχωρήσουμε προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τέτοια θέματα. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, είχαμε την ευκαιρία ε, να ξανακουβεντιάσουμε ορισμένα θέματα που έχουν σχέση με την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα των στατιστικών με τον αξιότιμο κύριο συνάδελφο που είναι και σήμερα εισηγητής και δεν θα χρειαστεί να επαναλάβω ορισμένες βασικές παρατηρήσεις. Από την προφορική παρουσίαση που μας έκανε ο εισηγητής μας κατάλαβα ότι τώρα και αυτό είναι περισσότερο υποψιασμένος τι κρύβονται πίσω από τα κείμενα και τις καλές διατυπώσεις όσο αφορά την αξιοπιστία και την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων. Δύο-τρεις παρατηρήσεις για να υπογραμμίσω το γεγονός ότι παρότι γίνεται μια προσπάθεια να εξασφαλιστεί καλύτερη ποιότητα στατιστικών στοιχείων, όσο αφορά την ύπαρξη πολιτικής βούλησης, και δεν απευθύνομαι στον εισηγητή μας, ξαναλέω ο οποίος ε, με βάση και την εμπειρία της προηγούμενης έκθεσης έχει, είναι πιο υποψεσμένος, Επιτρέψτε μου λοιπόν να αμφιβάλλω αν θα τα καταφέρει και αυτός ο κανονισμός να μας δώσει αυτό που θέλουμε. Και οι λόγοι είναι και εγγενείς. Ένας πρώτος λόγος, πολύ χοντρά το λέω, από τη στιγμή που η οικονομία και η κοινωνία καταγράφεται με αριθμούς και επομένως έτσι χαράζονται οι οικονομικές πολιτικές, κατά τη γνώμη μου υπάρχει μείζον πρόβλημα. Η στατιστική κατόπιν τούτου έχει την αξία της και έχει και την αξιοπιστία της. Μπορεί να λειτουργήσει για να κάνει σωστό σχεδιασμό, μπορεί να λειτουργήσει επικίνδυνα και να πάμε σε εξαπάτηση πολιτών. Το ερώτημα το δεύτερο είναι όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά με διάφορες καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί τι ζητάμε, τι στοιχεία ζητάμε και για ποια πράγματα. Και ανάλογα με το τι ζητάμε, ανάλογα αποτελέσματα πολλές φορές έχουμε που αποτυπώνει μια λυπή εικόνα μια κοινωνίας, μια οικονομίας και χαράζονται με συγκεκριμένε σκοπιμότητε πολιτικέ Υπάρχει πλούσια εμπειρία. Μιλάω, όπω ξέρετε, από την εμπειρία τη Ελλάδα, αλλά δεν είναι μόνο η Ελλάδα με τα Greek Statistics. Έχουμε αλλεπάλληλα τέτοια προβλήματα, απλώ βρέθηκε στην αιχμή του δόρατος, ε, διότι υπήρξαν εκεί τέτοια ζητήματα και επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί και ποινικά τα θέματα, το πώ καταγράφονται τα στατιστικά στοιχεία και επίσης δεν ξέρω πόσο η νέα οδηγία θα μας απαλλάξει από τη δημιουργική στατιστική. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο, θα κάνουμε και τις τροπολογίες, δύο-τρεις παρατηρήσεις επί της πιο συγκεκριμένης, ας το πούμε, προσπάθειας που γίνεται. Ποιος ελέγχει τις ανεξάρτητες αρχές. Εντάξει, να εξασφαλίσουμε την ανεξαρτησία. Ποιος την ελέγχει. Πώς το ελέγχουμε αυτό το πράγμα. Δηλα... Να σας πω, ξεκινώντας από την αρχή, ποιος ορίζει τον επικεφαλής της στατιστικής υπηρεσίας και με ποιο κριτήριο. Προφανώς θα είναι επιλογή κάποιου πολιτικού οργάνου κάποιας κυβέρνησης. Περνάει από κοινοβουλευτικό έλεγχο. Έχει μια ευρύτερη, ας το πούμε, καλή γνώμη. Τι σημαίνουν επαγγελματικά κριτήρια. Η εμπειρία περιορισμένη ενδεχομένω λέει ότι υπεύθυνο στατιστική υπηρεσία θα μπει ένα πρώην στέλεχο τράπεζα που η τράπεζα μπορεί να βαρύνεται και αυτή με όλες αυτές τις ιστορίες που μας στάσαν στην κρίση και μάλιστα μεγάλων τραπεζών ή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Διότι αυτή θεωρείται επαγγελματική εμπειρία. Αυτή η επαγγελματική εμπειρία εξασφαλίζει ότι ο επικεφαλής της στατιστικής υπηρεσίας έχει τα επαρκή επαγγελματικά κριτήρια, κατά μία έννοια έχει την αξιοπιστία ότι θα δουλέψει μόνος του, θα δουλέψει ανεξάρτητα. Αλλά το κρίσιμο ερώτημα, και τελειώνω εκεί θα δούμε και ότι... Ε, ποιος ελέγχει πόσο ανεξάρτητα αυτή η Επιτροπή δουλεύει. Ποιος έχει την πολιτική ευθύνη εν τέλει. Και τελειώνω με τη Eurostat. Θυμόσαστε ότι στην απόφαση της 26ης-27ης Οκτωβρίου του προηγούμενου χρόνου η Κομισιόν όρισε υπεύθυνο να παρακολουθεί το έργο της Eurostat τον κύριο Σεμέτα, τον αναγόρευσε και σε αντιπρόεδρο, είναι και αντιπρόεδρος. Στην ερώτηση αν κάνει κάτι στραβό η Eurostat, σκοπίμως στραβό, ποιος έχει την ευθύνη να το διορθώσει ή να πει αναλαμβάνω την ευθύνη. Τέτοια ερωτήματα υπάρχουν και δημιουργούν εύλογες, ε, εύλογες ενστάσεις. Αλλά δεν αναφέρομαι στον εισηγητή μας. Θα κάνει, ξέρω ότι θα κάνει φιλότιμη προσπάθεια και εμείς με τις τροπολογίες θα κοιτάξουμε να το βελτιώσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Uh, thank you very much. Uh, we have Mrs. From the... Σας ευχαριστούμε. Έχουμε από τη Eurostat έναν εκπρόσωπο, μία εκπρόσωπο μάλλον και θα ήθελε να κάνει κάποια σχόλια. Ίσως θέλετε να μας διευκρινίσετε κάποια πράγματα γιατί υπάρχουν ερωτήσεις και έχουμε λίγο καθυστερήσει. Παρακαλώ με μακρηγορήσετε. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Θα είμαι συνοπτικότατη, διότι νομίζω ότι πραγματικά ο ενθουσιασμός για την πρόταση και το αιτιολογικό που τη στηρίζει πολύ σωστά παρουσιάστηκαν από τον εισηγητή. Απλώς να αναφερθώ στην ακρόαση που έγινε με την παρουσία του κυρίου Ράντα του Γενικού Διευθυντή της Eurostat. Νομίζω η συζήτηση που επακολούθησε κάλυψε πολλά θέματα, τα οποία ούτως ή άλλως περιλαμβάνονται στις προτεραιότητες σας σήμερα. Η πρόταση κατά την άποψή μας είναι ιδιαίτερα ρεαλιστική. Τέτοιο επίπεδο φιλοδοξία σαφώ το χρειαζόμαστε και δικαιολογείται και από τα πρόσφατα επεισόδια που όλοι γνωρίζουμε. Είναι μια πρόταση που βρίσκεται στα όρια της επικουρικότητας. Είναι μια στοχευμένη αναθεώρηση και τα βασικότερα ζητήματα έχουν επεξηγηθεί με σαφήνεια. Απλώς τώρα θα ήθελα να σταθώ σε ερωτήσεις που τέθηκαν κατά την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε εδώ. Πρώτον, εάν οι ίδιες προδιαγραφές ανεξαρτησίας θα ισχύουν και για το Γενικό Διευθυντή της Eurostat. Η απάντησή μου είναι ναι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή προετοιμάζει μια αναθεωρημένη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ρόλο της Eurostat η οποία φροντίζει να υπάρξει πλήρη ευθυγράμμιση πρακτικών με τα όσα αναφέρει η πρόταση. Το δεύτερο σημείο αφορά τη δέσμευση, την εμπιστοσύνη, το σκοπό και τη διόρθωση της νέας αυτής πρότασης του ναυτοργαλείου. Βεβαίως πρόκειται εδώ για πολιτική δήλωση, αλλά αυτό που προέχει είναι η δήλωση πολιτικού χαρακτήρα και η ολοκλήρωση στην υλοποίηση να παρακολουθούνται, να ελέγχονται. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα καινοτόμο στοιχείο ώστε να μπορούμε να υπολογίζουμε στην επιβολή των όσων προβλέπει το κείμενο αυτό, να μην παραμένει δηλαδή κενό γράμμα στο χαρτί. Τώρα για την απέτηση για τα διοικητικά αρχεία και την πρόσβαση σε αυτά. Μας ενδιαφέρουν μόνο ποσοτικές πληροφορίες εδώ, μόνον ε, απλά δεδομένα. Αυτό θα πρέπει να το δούμε στο πλαίσιο τη μείωση του φόρτου εργασία και τη μείωση του κόστου. Δεν πρέπει να συλλέγουμε δεδομένα που ήδη υπάρχουν. Θέλουμε να αξιοποιούμε πλήρω τι διαθέσιμε πληροφορίε και συμφωνούμε βεβαίω ότι οι περιορισμοί χρειάζονται. Χρειάζονται, θα πρέπει να προβλεφθούν, διότι άλλα ζητήματα πέραν των ποσοτικών δεδομένων δεν μα ενδιαφέρουν. Ένα άλλο ε, ενδιαφέρον σημείο είναι η ανεξαρτησία έναντι της μεθοδολογίας και σε σχέση με τη μεθοδολογία. Κατά την άποψή μας είναι σημαντικό να υπάρχει μια σαφής συνένεση με τους χρήστες για το πώς θα χρησιμοποιούνται οι διάφορες έννοιες. Ευχαρίστως λοιπόν να συζητήσουμε στην απαρχή της διαδικασίας το θέμα αυτό, ώστε όσοι παράγουν στατιστικά δεδομένα να έχουν πλήρη ανεξαρτησία στην εφαρμογή της μεθοδολογίας τους, αλλά μια μεθοδολογία που να έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων. Αυτό νομίζω μπορεί να αποσαφινιστεί στο κείμενο. Φιλοδοξία μας δεν είναι να είμαστε απολύτως ανεξάρτητοι, Απλώ χρειάζεται μια σαφή συνένεση για τις διάφορες έννοιες και την μέθοδο. Σε ό,τι αφορά τον κώδικα πρακτικών, μιλάμε για ένα εργαλείο αυτορυθμιζόμενο. Μάλλον αν το εργαλείο της αυτορύθμισης είναι αρκετό. Θα πρέπει ο κώδικας πρακτικής να γίνει, να καταλάβουμε ότι είναι ένα κείμενο που θέτει ελάχιστα πρότυπα από τη μία. Αλλά προσπαθεί και να εμπνεύσει. Από αυτήν την άποψη λοιπόν είναι δύσκολο ένα τέτοιο εργαλείο να καταστεί απολύτως νομικό, νομικός δεσμευτικό. Η πρόταση αυτή προβλέπει κάποια ελάχιστα πρότυπα νομικώς δεσμευτικά, ιδίως έχουν να κάνουν με το πώς τα θεσμικά όργανα μπορούν να συμβάλλουν στην θέσπιση των στατικών αρχών, αλλά όχι κάτι άλλο ως προς τις διορθώσεις λόγου χάρη. Αυτά είναι τα βασικά σημεία στα οποία ήθελα να αντιδράσω σύντομα και απλώς να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει στην ενεργό στήριξη του Κοινοβουλίου προκειμένου να διαφυλάξουμε αυτό το επίπεδο φιλοδοξίας που έχετε και εσείς θέση. Θα πρέπει να παραμένει υψηλό το επίπεδο αυτό έως το τέλος της διαδικασίας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για τις συνεισφορές σας και Είμαστε πεπισμένοι ότι εδώ θα έχουμε μια εξαιρετική πρόταση που θα θέσει τα σωστά πρότυπα για την στατιστική και τον όλο ένα και σημαντικότερο ρόλο που διαδραματίζει στην κοινωνία μας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Πολλά η δουλειά έχει γίνει πρόσφατα για την στατιστική και γνωρίζουμε εκ πείρας ότι οι μάχες που δίνονται συνήθως έχουν αντιπάλους στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό πολλές φορές καταλήγουμε σε τριμερείς διαλόγους και για τη δική μου έκθεση υπάρχει ανεξελίξη ένα τέτοιο τριμερή διάλογο. Και στο πακέτο, στο, στη δέσμη μέτρων ε, για το Sixpack, ε, θελήσαμε να καλυφθεί η επαγγελματική ανεξαρτησία των στατιστικολόγων. Είναι ένα σημείο που μας ενδιαφέρει αυτό και θα πρέπει να το επιδιώξουμε. Προσπαθήσαμε να καταστεί αυτό ένα ορόσημο και στην έκθεση της κυρίας Φόρντ και θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία. Έντουαρτ. Ολοκληρώνοντας, να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδους εισηγητές, διότι πιστεύω ότι όλες οι παρατηρήσεις που ακούστηκαν ήταν χρήσιμες. Γίνεται μια σωστή διάκριση μεταξύ μιας έκθεσης που αντιμετωπίζεται απλώς ως ένα έγγραφο που θα πάρει την πορεία του και ενός εγγράφου με περιεχόμενο ουσίας που θέλει να επιφέρει πραγματικές αλλαγές. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τα σχόλια, ε, ιδίως για αυτά που αφορούν τα πρότυπα της Eurostat, το δεσμευτικό χαρακτήρα του κώδικα πρακτικών, το τι θα γίνει με τα διοικητικά αρχαία και τι ακριβώς εννοούμε με το σημείο αυτό, την ισορροπία μεταξύ ελευθερίας και ανεξαρτησίας ε, ταυτόχρονα, τι πολιτική κατεύθυνση θα πρέπει να δοθεί δηλαδή εδώ. Έπειτα, τελευταίο και πολύ σημαντικό, η πρόταση, η ποιότητα να απηχεί και την ρεαλιστική μέτρηση και καταμέτρηση. Να πω ότι έγινε ε, δήλωση στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη του ΟΣΑ ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να παρακολουθείτε ε, προσεκτικά με παράδειγμα τον δίκτυ για την ευζοία των οικογενειών λόγου χάρη. Να μην είναι ένα θεωρητικό θέμα, αλλά να παρακολουθείτε το βιωτικό επίπεδο των οικογενειών στην πράξη λόγου χάρη. Θα σταθώ εδώ και στις αρχές Σεπτεμβρίου θα παρουσιάσω και τις ε, τροπολογίες για την έκθεση αυτή. Σας ευχαριστούμε προσωρινό χρονοδιάγραμμα. Παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης στην Επιτροπή στις 26 Σεπτεμβρίου με προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών στις 9 Οκτωβρίου. Θα εξεταστούν στις 5 Νοεμβρίου και θα ψηφίσουμε στις 28 του μήνα. Ενδεχομένω να περάσει το θέμα αυτό από τον Ολομέλεια τον Δεκέμβριο. Ίσως και λίγο νωρίτερα, αλλά μάλλον τον Δεκέμβριο. Τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε. Σημείο 8. Ψηφοφορίες. Αναβάλλεται η ψηφοφορία για τη MIFID, οπότε θα ψηφίσουμε μόνο για το κοινό σύστημα φορολόγηση των τόκων και των δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιριών διαφορετικών κρατών μελών. Θα σας δώσω ένα δίλεπτο να βεβαιωθείτε ότι έχετε όλοι τους καταλόγους σας. Yeah, okay. Yeah, it's okay. But people are still Are we, are we ready? Um, let's... Είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πιέσατε το κομβίον παρακαλώ. Okay, um... oh, yes, you see No. Right, 35 35 βουλευτές έχουν βάλει την κάρτα, 5 δεν έχουν ψηφίσει ακόμα. Κύριε Κλίντς, έχω ξεχάσει την κάρτα μου η απάντηση, οπότε μείον ένας από τους ε, φιλελεύθερους. 36 κάρτες στην υποδοχή, 31 έχουν ψηφίσει. Δύο από τους φιλελεύθερους. Εξαρτάται. Λοιπόν, πέρας της ε, ψηφοφορίας. Ξεκινάμε λοιπόν. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 15 δεν ψηφίζεται μάλιστα. 4 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε τη 17. Μπορείτε να ξεκινήσετε την ψηφοφορία. Ωραία. Συν ε, δύο που έχουν ε, να προσθεθούν από την Άλντε υπέρ. Λοιπόν, πέρας. Άρα είναι 20 υπέρ, 17 κατά. Οπότε δεκτή. 18 υπέρ, κατά. Αποχές Νομίζω πως είναι δεκτή με παρόμοια πλειοψηφία όπως πριν. Να την επαληθεύσουμε όμως. Ψήφισαν όλοι, συν άλλοι δύο από τους φιλελεύθερους, οπότε έχουμε 21 υπέρ, 16 κατά, δεκτή. 19 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Νομίζω παρόμοια όπως πριν. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Χωριστή ψηφοφορία για την 21. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Μέρος δεύτερον υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ναι. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 6 υπέρ. Όχι. Να, με συγχωρείτε. 23 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 24 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 7 έχει καταπέσει. 25 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 1 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Σε τρία μέρη η 8. Μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτή να την επαληθεύσουμε. μου μοιάζει με την ίδια συμπεριφορά. Συν δύο να προσθέσουμε από τους φιλελεύθερους. Κάποιος άλλος να ψηφίσει όχι πέρας. 20 υπέρ, 17 κατά με τους δύο συναδέλφους από την άλλη. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές δεκτή η ίδια πλειοψηφία. Μέρος τρίτο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές δεκτή. 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τώρα ηλεκτρονικά ψηφίζουμε το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 32 υπέρ. 3 κατά και 3 αποχές. Επί του νομοθετικού ψηφίσματος τώρα άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι κατατίστε το κουμπί πατημένο. Ευχαριστώ. Πέρας. 33 υπέρ. Μία κατά τρεις αποχές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω πως λύεται η συνεδρίαση. Όχι. Ναι, ναι, μέχρι το απόγευμα. Διακόπτεται. He's not here, is he? Oh, oh, I'm sorry, I couldn't see Um, sorry, I, I think did the rapporteur wish to make Για την αναβολή της προφορίας της οδηγίας MIFID. Αναβολή είναι, μας ενημερώνει ο εισηγητής, επειδή απλώς είναι πάρα πολύ σοφόρτος και αναβλήθηκε.